συζήτησης η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις επιτρεπόμενες διαστάσεις και το βάρος ορισμένων οδικών οχημάτων. Και θέλω πρώτα να δώσω το λόγο στον συντάκτη της προφορικής ερώτησης, τον κύριο Σίμψον, για πέντε λεπτά. Uh, Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματο τη Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ζήτησα να συζητηθεί απόψε το ζήτημα των βάρου ε, και των διαστάσεων για τα λεγόμενα γιγαντιαία φορτηγά. Μετά από μια ερώτηση που ετέθη πέρσι για το δικαίωμα της Κομισιόν να ανασυντάξει μονομερός την νομοθεσία για τα γιγάντια φορτηγά χωρίς να συμβουλευτεί τους συνομοθέτες. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ της επέκτασης της χρήσης αυτών των φορτηγών γιατί θεωρώ πως οι υποδομές σε πολλές χώρες δεν μπορούν να τα υποδεχτούν και έχουμε ζητήματα οδικής ασφάλειας και βεβαίως υπάρχει και δεν υπάρχει αξιολόγηση της απειλής στο περιβάλλον και στον τομέα των σιδηροδρόμων. Τώρα, είτε υπέρ είναι κανείς είτε κατά, η Επιτροπή μας συμφωνεί πως οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της συναπόφασης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πως κάτι τόσο σημαντικό μπορεί να αποφασιστεί με τρόπο αυθαίρετο, να ανακοινωθεί σε κάποια διάσκεψη με βάση του ότι κάποιος εκεί πέρα νομικός αποφάσισε να αλλάξει την απόψή του. Μας είπανε στο παρελθόν πως πως ε, δεν μπορεί να υπάρξει παράταση με απόφαση μόνο της Κομισιόν και αυτό μάλιστα μετά από ερώτηση βουλευτή. Και μετά ως διαμαγείας η πρόθεση της Κομισιόν ήταν να το περάσει κρυφά mm. και ε, ήλπιζε πως δεν θα το προσέξει το Κοινοβούλιο. Το πρόσεξε όμως κυρία Πρόεδρε και είχαμε μετά μια φαρσοκομωδία. Η Κομισιόν κρύβεται, προσπαθεί να φύγει από το, να ξεφύγει από την κατάσταση την οποία δημιουργήσε. Μετά από μήνες περίσκεψης η Κομισιόν αποφάσισε και ο Επίτροπος συγκεκριμένα να επιμείνει στην ε, νέα του ερμηνεία. Παρά το ότι παραδέχθηκε σε επιστολή προς τα εμένα πως δεν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και ακόμα και ο πρόεδρος Μπαρόζος, επιτροπή προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον ε, κύριο Σούλτς, παραδέχτηκε πως δεν δημιουργείται απόλυτη νομική βεβαιότητα. Ζητώ λοιπόν απόψε από τον κύριο Επίτροπο να συμφωνήσει μαζί μου πως η νομοθεσία είναι ασαφής και πως υπ' αυτές τις συνθήκες έχει καθήκον να δώσει τέλος στην ασάφεια με το να υποβάλει προς το Κοινοβούλιο για εξέταση αναθεώρηση της νομοθεσίας που θα βλέπει τα ζητήματα της διασυνοριακής κυκλοφορίας γιγάντιων φορτηγών. Μου λένε πως δεν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο και έτσι εδραιώνονται τα περσινά λάθη. Εάν η επιθυμία σας είναι να επεκταθεί η χρήση αυτών των φορτηγών, τότε καλά θα κάνετε να έχετε το θάρρος της γνώμης σας να φέρετε αυτές τις αλλαγές στο Κοινοβούλιο υπό την απόφαση για να τις εξετάσουμε με τρόπο δημοκρατικό. Χρειάζεται εδώ πέρα νομική σαφήνεια, κύριε Επίτροπε, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πλήρη συνεργασία του συνομοθέτη και όχι επειδή έτσι κάπνισε σε κάποιον δικηγόρο στην Κομισιόν. Το όλο ζήτημα έχει γίνει πλέον ένα χάλι και μισό, το δημιούργησε η Κομισιόν και θα πρέπει να το λύσει με το να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να παίξει τον θεσμικό του ρόλο όπως αυτός περιγράφεται στις συνθήκες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σίμψον τώρα ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επιτροπό Κάλλας, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Κομισιόν ε, ευχαριστεί τα μέλη τη Επιτροπή Μεταφορών για την ευκαιρία να συνεχιστεί η συζήτηση για την αναθεώρηση της οδηγίας 96 53 ΕΚ η χρήσιμη συζήτηση που έλαβε χώρα από την άνοιξη του 2012 τόνισε ότι είναι λεπτό το θέμα αυτών των μακρών φορταγών και των διαφορετικών ερμηνεών που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τη μεταχείρισή του δύναμη τη οδηγία. Επίση, επιβεβαίωσε ότι χρειαζόταν διευκρινήσει για τα θέματα αυτά. Η Κομισιόν ολοκληρώνει την αναθεώρηση της οδηγίας. Ε, μία πρόταση μπορείτε να την αναμένετε τον επόμενο μήνα και θα ακολουθεί η τακτική νομοθετική διαδικασία. Χρειάζεται η αναθεώρηση να προσαρμόσει την οδηγία στις τεχνικές εξελίξεις και ε, στις, ε, στις οικονομικές και κοινωνικές επιτακτικές ανάγκες, κυρίως για τις διατροπικές μεταφορές. Θα επικεντρωθεί σε αλλαγές που θα φέρουν σημαντικά ωφέλη, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη σύνδεση μεταξύ τρόπων μεταφορών, καθώς και την επιβολή του νόμου αυτές οι αλλαγές καταρχήν θα ε, επιτρέψουν την αερονομικό streamlining των οχημάτων ε, και θα καθοριστούν τεχνικές απαιτήσει ε, και για τα FE φορτηγά. Επίσης θα διευκολυνθεί η μεταφορά των κοντέινερ 45 ιντσών στην διατροπική μεταφορά. Τρίτον, θα προσαρμοστεί το μέγιστο βάρος για να προθεθεί η χρήση ε, κάποιων καθαρών συστημάτων όθησης των ε, ηλεκτρικών μηχανών και θα υπάρξουν διατάξεις για την επιβολή, για τη μείωση ε, της υπερβολικής φόρτωσης του overloading και επίσης για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση για τη διασυνοριακή κυκλοφορία των, ε, μακρό, των μεγάλων φορτηγών. Αυτά τα θέματα μπορεί να συζητηθούν ε, στα πλαίσια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας που σχετίζεται με αυτή την οδηγία. Έτσι λοιπόν ε, σεβόμαστε πλήρως την άποψη της Επιτροπής, την γνωμοδότηση της Επιτροπής για το θέμα αυτό και θα ακολουθήσουμε την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για τη συνεχιζόμενη συζήτηση μεταξύ των δύο οργάνων και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η επικοδομητική συνεργασία όταν η πρόθεση αναθεώρησης της οδηγίας 96 53 ΕΚ θα έχει θετηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Κάλλα. Και τώρα να περάσουμε στου ομιλητέ εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Καταρχήν εκ μέρου του ΕΛΚ, ο κύριο Μπαχ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Κάλλας, πολλές φορές ανακοινώσατε μια μεταρρύθμιση της οδηγίας 96-53 όσον αφορά τις επιτρεπόμενες διαστάσεις και το βάρος κάποιων οδικών οχημάτων. Και αναφερθήκατε σε κάποια άλλα ζητήματα όπως βελτίωση της αεροδυναμικής και ασφάλειας των οχημάτων, ε, περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη και προσαρμογή των οχημάτων στις απαιτήσεις σύγχρονης τεχνολογίας. Το ερώτημά μου στο πλαίσιο αυτό είναι θα ασχοληθεί η Κομισιόν με αυτό το οποίο ανακοινώσατε εσείς τον Ιούνιο κύριε Κάλλας ε, και το υποσχεθήκατε σε επιστολή του Προέδρου Μπαρόζο δηλαδή να δημιουργηθεί σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου ε, όσον αφορά τα λεγόμενα γιγαντιαία φορτηγά, τα υπερμεγέθη αυτά φορτηγά. Κάποια κράτη-μέλη είχαν κάποιες θετικές εμπειρίες, κάποια άλλα λιγότερο θετικές ε, και κάποια άλλα αναστέλουν την χρήση τους. Τα προβλήματα είναι γνωστό, δεν υπάρχουν οδικές υποδομές και δεν έχουν ξεκαθαρίσει ζητήματα οδικής ασφάλειας και επίσης δεν συμβάζονται αυτά με το σκεπτικό να πάει περισσότερη κυκλοφορία από τους δρόμους στους σιδηρόδρομους ε, και άλλα ζητήματα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Οπότε συμφωνώ πλήρω με τον πρόεδρό μα, τον κύριο Μπράιν Σίμψον. Γνωρίζετε τη θέση του Κοινοβουλίου και θα επιθυμούσα να κινηθείτε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να έχουμε μια συνεκτική θέση και στο πλαίσιο ε, της επανεξέτασης θα μπορούσαμε να δούμε παραδείγματος χάρη τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, και των υφιστάμενων δυνατοτήτων. Μόνο με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια λογική νομοθεσία. Η μονομερή ερμηνεία από πλευράς κομισιών τελικά δεν βοηθάει κανέναν ούτε ε, το κυκλόφωνος στον δρόμο, ούτε τον κλάδο. Σας ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Αλχαντραουή. Ευχαριστώ. κυρία κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν αντιλαμβάνουμε από την απάντηση του Επιτρόπου το τι ισχύει ακριβώς. Εμείς λοιπόν ανησυχούμε για το θέμα αυτό πρώτα απ' όλα για τους λόγους της διαδικασίας αλλά βεβαίως και για το ζήτημα της ε, ουσίας. Όσον αφορά την ε, διαδικασία μας εκπλήσει το ότι η Κομισιόν μονομερός οδηγήθηκε σε δική της ερμηνεία για ένα ζήτημα ε, κρίσιμα, κρίσιμο όπως τα υπερμεγέθη αυτά φορτικά Και βεβαίω δεν είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα διαστάσεων και βάρους και εφόσον ξεκαθαρίστηκε από τις ερωτήσεις των ε, συναδέλφων πως δεν ήταν αυτό το ζήτημα πλέον δεν μιλάμε για κάποιο λεπτομεριακό ζήτημα αλλά για ζήτημα νομοθεσίας αλλά βεβαίως όταν ξέρουμε μεταξύ, ποιο είναι το καθεστώς της υφιστάμενης ε, νομοθεσίας. Εμείς θέλουμε λοιπόν μια δημοκρατική συζήτηση και ζητάμε την δική σας συμμετοχή. Δεύτερον, επί της ουσίας, ε, το να ενθαρρύνουμε τα όλο και μεγαλύτερα φορτηγά αντιβαίνει σε αυτό το οποίο λέμε στη Λευκή Βίβλο για το ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε ειδικά στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων σε μεγαλύτερη χρήση των σιδηροδρόμων. Για όλους αυτούς τους λόγους σας ζητάμε να μην προχωρήσετε με τα σχέδιά σας και να ασχοληθείτε με άλλα πιο σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ για τους ε, φιλελεύθερους κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλάμε για μια οδηγία η οποία είχε συνταχθεί σε καιρούς διαφορετικούς όταν δεν ήταν τόσο πολύ καιρό τα φορτηγά στο δρόμο. Και μην ξεχνάμε πως ε, μετά προσθέθηκαν άλλες χώρες οι οποίες μετά άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Και τι γίνεται. Εδώ πέρα μας ε, μας λέει η Κομισιόν πως ε, κάτι τέτοιο είναι προς το Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να μάθουμε ποια είναι η υφιστάμενη νομική κατάσταση. Επιτρέπεται αυτά τα φορτηγά να διασχίζουν τα σύνορα. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι και ιδεολογικό, αν αρέσουν σε κάποιον ή όχι. Εγώ, εμεί στην Κάτω Σαξονία είχαμε θετικέ εμπειρίε με αυτά, αλλά το ζήτημα είναι εάν επιτρέπεται να διασχίζουν τα σύνορα ή όχι. Και ακριβώ το πρόβλημα εδώ πέρα είναι πω η Κομισιόν έχει δώσει διαφορετικέ απαντήσει. Πρώτα απ' όλα σε μία ερώτηση απαντα... δόθηκε απάντηση πω δεν επιτρέπεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Και πως ε, αν γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να δίνεται ειδοποίηση. Μετά ε, ο ίδιος ο Επίτροπος ο κύριος Κάλλας είπε πως ε, δεν βλέπουμε πώς ε, μπορεί να απαγορευτεί το να διασχίσουν τα σύνορα. Εμείς το επιτρέπουμε στην κάτω Σαξονία. Η Ολλανδία επίσης και μας είπε ο κύριος Κάλλας πως δεν είναι δυνατόν και λογικό να σταματάνε στα σύνορα. Οπότε το θέμα είναι, κατά την άποψή μας, είναι πως οι επιχειρηματίε πρέπει να έχουν μια νομική ασφάλεια. Επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα φορτηγά αυτά. Ε, και ίσως, ξέρετε, να μην έχει καμία λογική να μην τα χρησιμοποιούν ε, ε, αν δεν είναι εκτός συνόρων. Οπότε πρέπει να ξεχαρίσει η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση για να έχουν και νομική ασφάλεια επιχειρήσει. Σα ευχαριστώ για του πράσινου, Ο κύριος Κράμερ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ο Κόνραντ Αντενάουερ είχε πει όταν άλλαξε ξαφνικά άποψη πως καμία δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να με εμποδίσει να γίνω εκ των υστέρων εξυπνότερος. Το ίδιο ισχύει και για τον Επίτροπο. Το Μάρτιο του 2010 όταν του είχα απευθύνει μια ερώτηση σχετική είχε απαντήσει ξεκάθαρα όχι και είπε πως ε, εάν η Κομισιόν ε, μάθαινε για διασυνοριακή χρήση τέτοιων φορτηγών θα κινούσε διαδικασία επί παραβάση κατά του κρατσμέλους. Και όταν τον ε, ρώτησε η International Road Union για το ίδιο θέμα, έδωσε τελείως διαφορετική απάντηση και έλεγε βεβαίως δεν υπήρξε καμία αλλαγή, απλά διαφορετική ερμηνεία του νόμου. Ξαφνικά ο θεματοφύλακας των συνθήκων παραβίαζε τον νόμο. Αυτό εξόργησε όλες τις ε, ομάδες ανεξαρτήτως του αν ήταν υπέρ ή κατά των φορτηγών αυτών. Την δε Ιούνιο του 2012 ο κύριος Κάλλας είπε πως θεωρώ πως δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα παρά το ότι δεν είναι ξεκάθαρη εντελώς αυτή η γραμμή. Και για να ξεκαθαρίσει κάθε αμφιβολία όσον αφορά την ε, κατάσταση μίλησε για αναθεώρηση της οδηγίας την οποία ανέφερε ο πρόεδρος Μπαρόζο όταν τον ρώτησε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και του, σχετικά και του ζήτησε να σταματήσει ο αρμόδιος επίτροπος αυτές τις ε, έκνομες πρακτικές. Αλλά και σε συνέντευξη στο Europolitics ο κύριος Κάλλας είπε πως ε, θα υπάρξει μια αναθεώρηση αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα στα σχέδιά μας. Ε, νομίζω πως μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το οποίο πει ο Αντενάου στην περίπτωσή σας και να πει πως καμία δύναμη του κόσμου δεν μπορεί να με εμποδίσει να γίνω πιο χαζός εκ των υστέρων. Σας ευχαριστώ. Έχετε μία μπλε κάρτα από την κυρία Μάισνερ. Θα έχετε την ερώτηση, ναι. Κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Ναι, ο κύριος ε, Κράμερ ε, βεβαίως ε, μίλησε για βλακεία του Επιτρόπου και τον κατηγόρησε για σοβαρά πράγματα. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να παραμείνουμε στην ουσία της συζήτησης. Ε, το ερώτημά μου συγκεκριμένα. Μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα όντως για παραβίαση του νόμου όταν δεν είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν και είναι απόφαση των κρατών μελών την οποία απλά κοινοποιούν στην Κομισιόν. Άρα για ποια παραβίαση μιλάμε. Η Κομισιόν απλά λαμβάνει γνώση. Ναι κύριε Κράμερ. Πριν από δύο χρόνια ρώτησα ρητός τον Επίτροπο εάν γνωρίζει για την, ε, το εάν επιτρέπεται αυτά τα φορτηγά να διασχίζουν το σύνορο. μου είπε ρητός όχι. Και συμπλήρωσε την απάντηση και είπε και αν μάθω κάτι τέτοιο, αν επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο τα κράτη-μέλη, θα ζητήσω να το σταματήσουν και αν δεν το κάνουν θα κινήσω διαδικασία επί παραβάσεις, βάρος του κράτους. Εμπιστεύτηκα εγώ τον Επίτροπο. Και ξαφνικά μου λέει, μα ε, τώρα το ερμηνεύω αλλιώ. Εγώ κρίνω πώς ερμηνεύονται οι νόμοι, δεν με ενδιαφέρει το Συμβούλιο, δεν με ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Mm. Ε, δεν είναι δημοκρατία αυτό. Και γι' αυτό συμφωνήσαμε όλες οι ομάδες στην Επιτροπή ότι δεν είναι πράγματα αυτά, δεν μπορεί να παραμερίζουν το Κοινοβούλιο, πρέπει να υπάρξει νομοθετική διαδικασία. Σταματήστε τι παρανομίε μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, ήσασταν άτυχος τελευταία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχατε το πακέτο των αεροδρομίων που απορρίφθηκαν οι προτάσεις σας. Και τώρα έχω την υποψία πως ε, έχετε την εξή αίσθηση. Άμα δεν κάνουν αυτό που θέλω, δεν θα ασχοληθώ μαζί τους. Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό κάνετε εδώ πέρα με τα φορτηγά. Μας λέτε ε, για βάρο και διαστάσεις και αυτό δεν έχει σχέση με την ουσία του ζητήματο. Εδώ πέρα έχει δίκιο ο κύριο Κράμερ. Από μόνο σα. και πιθανώ χωρίς νομιμοποίηση αλλάξατε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν γίνονται αυτά κύριε Επίτροπε. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι, πρέπει να υποβάλλετε νομοθετική πρόταση. Αλλιώς δεν κάνετε τίποτα. Θέλω να σας ρωτήσω. Θέλετε να είστε ο πρώτος Ευρωπαίος Επίτροπος στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει κάτι αντίστα με τη βούληση του νομοθέτη. Δεν νομίζω να είναι αυτή η πρόθεσή σας. Αλλά προς τα εκεί οδεύετε. Κύριε Επίτροπε, ε, σας άκουσα στην ε, τοποθέτησή σας ε, σε αυτά τα οποία πατήσατε στον κύριο Σίμψον και είπατε πως γνωρίζετε πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα. Ε, προφανώς δεν το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, άμα δείτε το τι έχετε κάνει τους τελευταίους μήνες, προφανώς δεν αντιλαμβάνεστε την ευαισθησία του ε, ζητήματος και αν τίθεται κάτι ένα αμφιβόλο, σας ενδιαφέρει μόνο ένα συγκεκριμένο τομέα. Σας άκουσα, μιλήστε για αεροδυναμική, ε, βάρος, διαστάσεις, προσαρμογή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ε, δηλαδή, καταλαβαίνω, θέλετε να αποφύγετε την υπερβολική φόρτωση με το να αυξήσετε τόσο πολύ το όριο του βάρους που να μην είναι δυνατόν να μιλήσουμε για υπερφόρτωση να μην έχει καμία ευκαιρία ο σιδηρόδρομος πλέον να είναι ανταγωνιστικός. Το ερώτημά μου είναι, θα κάνετε πραγματική αξιολόγηση αντικτύπου που θα βλέπει και το επιπρόσθετο κόστος για το δημόσιο τομέα εάν επιτραπούν αυτά τα φορτηγά στους δρόμους μας. Σας προειδοποιώ, οι Άλπεις θα αντισταθούν. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Κάλλας, επανειλημμένως έχει πει ότι είτε στα τέλη του 12 είτε στις αρχές του 2013 θα να εφαρμόσει την οδηγία 996 που καθορίζει ότι τα διάφορα οχήματα που κυκλοφορούν του τρόμου της Ένωσης θα έχουν ανώτατες διαστάσεις και εθνικός και διεθνός με προκαθορισμένο τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή το ΕΡΚ και το Συμβούλιο πρέπει να τα ξαναδούνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συγχωρείτε, και το Συμβούλιο. Γιατί αυτή τη στιγμή συζητιούνται τα θέματα των ψηφιακών ταχογράφων, ταχυγράφων και εμείς πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή του μηχανήματος αυτού θα έχουμε χρήσιμες πληροφορίες και για τις ε, διαδικασίες φόρτωσης-εκφόρτωσης και άρα στο Συμβούλιο μας είπαν, η Επιτροπή δήλωσε προς το Συμβούλιο ότι θα αλλάξουν όλα αυτά, γι' αυτό σας ερωτώ κύριε Επίτροπε άμεσα. Η τροποποίηση της οδηγίας 53 θα έχει μέσα τον ταχογράφο ή όχι τον ταχυγράφο. τον κύριο Ερτούκ. τώρα η οφθαλμοθυρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, σήμερα το απόγευμα μετά από 9 εβδομάδες έλαβα απάντηση στο ερώτημά μου. Σύμφωνα με το άρθρο 170 ε, έχει 6 εβδομάδες περιθώριο η Κομισιόν απαντήσει, αλλά αυτό τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Μου είπατε ξεκάθαρα πώς επιμένετε στην νέα σας ερμηνεία. Και σας λέω ξεκάθαρα πως αυτή η διαδικασία είναι απαράδεκτη, κύριε Επίτροπε, η νέα αυτή ερμηνεία καταργεί την διάκριση των εξουσιών από την πίσω πόρτα. Πρέπει να υποβάλλετε πρόταση στην τακτική νομοθετική διαδικασία ενώπιον του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αλλαγή της οδηγίας 9653 αλλά θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση ειδικά για τη διασυνοριακή κυκλοφορία. Εκεί πέρα ακριβώς είναι το ζήτημα και αυτή ήταν η πρόθεσή σας. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ερτούκ. Συνάδελφος Κράμερ θέλει να σας θέσει μια ερώτηση. Δέχεστε. Να ρωτήσω τον κύριο Ερτούγ εάν γνωρίζει αν διασχίζουν κάπου τα σύνορα αυτά τα φορτηγά και τι σκοπεύει να κάνει. Και θα ήθελα να ε, ζητήσω τον κύριο Επίτροπο να τοποθετηθεί για αυτές τις παρανομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ερτούγου. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Σημαντικό ερώτημα. Πράγματι, από όσο γνωρίζουμε, σήμερα τέτοια φορτηγά πηγαίνουν μεταξύ Δανίας και Γερμανίας. Και εδώ είναι το ερώτημα προς εσάς. Πότε σκοπεύετε κύριε Επίτροπε ως ε, θεματοφύλακα στο συνδικό να κινήσετε διαδικασία επί κατά των δύο αυτών χωρών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Έρτου. Ο κύριος, η κυρία Αγιάλα Σέντε ζήτησε το λόγο επίσης στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, με αυτή τη σύγχυση που προκαλείται, κύριε Επίτροπε, ε, στη χώρα μου, στην Καταλωνία μόλις διατήθηκε ε, ένας ε, κανόνας για 300.000 τόνους ακριβώς για ε, λόγω αυτής της σύγχυσης επειδή δεν ξέρουμε πώς να ερμηνεύσουμε την νομοθεσία. Εγώ νομίζω ότι ε, δεν υπάρχει ασφαλή δικαίωση, δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ξεκαθαριστεί το συντομότερο αυτή η κατάσταση και για να, δημιουργούνται, ε, να μην δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών. Πρόεδρος, ευχαριστώ τη συνάδελφο Αγιάλα Σέντερ. Κύριε Κάλλας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εξότιμα μέλη. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχουμε κάνει πολλά και σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι τόσο μεγάλη λοιπόν η σύγχυση. Η Κομισιόν ε, δεν έχει καμία πρόθεση να ε, δώσει την άδεια να χρησιμοποιούνται αυτά τα πολύ μεγάλα φορτηγά παντού στην Ευρώπη. Ε, εγώ υποστηρίζω ότι αυτό πρέπει να ρυθμίσετε από τα κράτη-μέλη αν τα κρατή-μέλη επιτρέπουν σε αυτά τα μεγάλα φορτηγά να χρησιμοποιούνται, όπως συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες, τότε αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αν ε, υπάρχουν χώρες ε, των οποίων ο πληθυσμό δεν αρέσκεται να χρησιμοποιούνται αυτά τα μεγάλα φορτηγά, τότε μπορούν οι χώρες να αποφασίσουν να τα απαγορεύσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσετε το θέμα. Εμείς δεν έχουμε την πρόθεση να επιτρέψουμε τη χρήση αυτών ε, των φορτηγών σε όλα τα κράτη-μέλη. Ήθελα να πω ότι αυτή η τροποποίηση της οδηγίας συμπεριλαμβάνει πολλές θετικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις και το βάρος για να έχουμε φορτηγά πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικά. Γι' αυτό το ανέφερα αυτό στην αρχή. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ορισμένα κράτη-μέλη επέτρεψαν να κυκλοφορούν αυτά τα μεγάλα φορτηγά και το ίδιο ισχύει και για πολλά κρατηδία στη Γερμανία. Υπάρχουν διάφορες ε, εκθέσεις, ε, κάποιες εκθέσεις ε, λένε, κάποιες αναφορές λένε ότι είχαμε μελέτη που και εξυλογήσαμε τρόπο την κατάσταση και όπως είπε και ο κύριος Μπαχ, Υπάρχουν πολλαπλές απαντήσεις ε, σε αυτά τα ερωτήματα. Τώρα, για το αν ήταν αντικρώμενη η δική μας άποψη και αν δημιουργήθηκε έτσι πρόβλημα, παραδέχομαι ότι αυτό ήταν ένα λάθος να δοθεί μια νομική απάντηση σε μια επιστολή, ή σε ποια είναι η νομική ερμηνεία και θεωρούμε ότι αυτό αρκεί. Αν ε, διαβουλευτήκαμε και με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και όπω γνωρίζετε, ήταν όλα τα μέλη τη Επιτροπή Μεταφορών παρόντα να συζητήσαμε αυτό το θέμα, ότι αρκεί αν δώσουμε νομικέ εξηγήσει και αν οι χώρε επιτρέπουν τη χρήση μεγαλύτερων φορτηγών, μπορούν αυτά να περάσουν και τα σύνορα αν πληρούνται ορισμένε συνθήκε. Και οι συνθήκε αυτέ ε, αναφέρονται στον κατάλογο. Και συμφωνώ ότι φυσικά ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Παραδέχομαι ότι ήταν λάθος παραδέχομαι ότι ήταν δικό μας λάθος και θα μπορούσαμε να το έχουμε διαχειριστεί, να το έχουμε αντιμετωπίσει δύναμη αυτής της οδηγίας. Τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι λοιπόν, το Κοινοβούλιο έχει πλήρη αρμοδιότητα για να προτείνει οποιαδήποτε τροπολογία στην οδηγία αυτή. Επομένως θα ρυθμιστεί το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Είναι τώρα στα χέρια της Επιτροπής Μεταφορών να γνωμοδοτήσει για τις δυνατότητες αυτές, ε, για την ε, διασυνοριακή διέλευση των φορτηγών. Υπάρχει νομική εξήγηση μέχρι τώρα. Η νομική μας άποψη είναι ότι αν επιτρέπουν τα κράτη-μέλη αυτά τα μεγάλα φορτηγά να χρησιμοποιούνται να κυκλοφορούν, ότι μπορούν και αυτά να περάσουν τα σύνορα. Εμείς ε, διστάσαμε να συμπεριλάβουμε ε, τεχνογράφηση αυτή την οδηγία γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά μηχανήματα και προωθούμε την ε, εθελοντική χρήση αυτών των αισθητήρων. Δεν ε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιβαραβάση κατά 100 κρατών μελών που έχουν ε, επιτρέψει σε αυτά τα μεγάλα φορτηγά να περάσουν τα σύνορα. Σας ευχαριστώ. Now. Dear colleagues, the discussion has been... Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Ο Επίτροπος υποθέτω πως θα είναι στη διάθεσή σας μετά το τέλος της συνεδρίασης, εάν επιθυμείτε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις ε, παρεμβάσεις σας. Σας ενημερώνω πως η συνεδρία θα επαναληφθεί αύριο το πρωί σε 9. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.